Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρία. Είναι κοινή συνεδρίαση τη οικονομική Επιτροπή και χαιρετίζω τον πρόεδρο αυτή τον κύριο Γκαλτιέρη, και τη Επιτροπή Tax 2 που αποκαλείται για τα φορολογικά. Είμαι ευτυχή που σα παρουσιάζω τώρα. Μάλλον σα δίνω τι καλύτερε ευχές για τον καινούριο χρόνο. Ελπίζω ο νέο χρόνο να είναι καλύτερο από τον προηγούμενο και σίγουρα θα είναι επιφορτισμένος όσον αφορά τις επιτροπές μας. Έχουμε πολλή δουλειά. Θα είδατε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Αν έχετε, δεν έχετε παρατηρήσεις, υιοθετείτε ένα σημείο που είναι ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο, τον κύριο Μοσκοβισή. Έχετε στο φάκελό σας τις διαθέσιμες γλώσσες. Η συνεδρίαση αυτή, όπως και όλες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής ΤΑΞ, είναι δημόσια ανοιχτή συνεδρίαση και μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Μαζί με τον πρόεδρο Γκουαλτιέρη και σε συμφωνία με τον Επίτροπο που χαιρετίζω και τον ευχαριστώ που ήρθε εδώ, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά και τις εργασίες της Επιτροπής TAX 2 που παρατείνει τις εργασίες της προσωρινής Επιτροπής TAX 1 ακούγοντας τον Επίτροπο που είναι φορτισμένος σε φορολογικά θέματα, ώστε να μας ενημερώσει να μας ανακοινώσει τα αποφασιστέντα της περασμένης εβδομάδας όσον αφορά την υλοποίηση διαφορών μέτρων και αυτά που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επόμενες εβδομάδες. Να επενθυμίσω ότι η TAX 2, η Επιτροπή αυτή, έχει λάβει εντολή. Θα παρακολουθεί τα όσα έχουμε κάνει και γίνονται στην Επιτροπή και έγιναν στην Επιτροπή TAX 1 να ολοκληρωθεί η συλλογή των πληροφοριών, με άλλα λόγια, των πληροφοριών που δεν συνελέγησαν άπασες, όπως στο, στην ομάδα του Διευθυντικού κώδικα, το γνωρίζει πολύ καλά αυτό το θέμα ο Επίτροπος ο κ. και θα μας ενημερώσει δεόντως Θέλουμε να ολοκληρώσουμε και τις ακροάσεις που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε στην πρώτη φάση και κυρίως η έντολή μας αφορά την εποπτεία υλοποίηση των συστάσεων που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την έκθεση της ΤΑΞ και της Επιτροπής της Οικονομικής και κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί όλες οι αποφάσεις και στο Συμβούλιο Υπουργών και στα κράτη-μέλη και στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο που εφαρμόζονται του ΩΣΑ. Στα πλαίσια του ΤΑΞ 1 διαπιστώσαμε εκ νέου τη σημασία που έχει η φόρο διαφυγή που πραγματοποιούν διάφορες πολυεθνικές εταιρείες και έχουμε την εντύπωση ότι άρχισε να αλλάζει η νοτροπία χάρη στη συνδυασμένη δράση των Επιτροπών του Κοινοβουλίου και του ΩΣΑ. Και θέλουμε να ξέρουμε κύριε Επίτροπε, τώρα στις αρχές του έτους, τι πρωτοβουλίες νέες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά αφορά αυτά τα θέματα και ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ αλλά και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μοσκοβισή Πού παρίσταται. Ευχαριστώ αλλά για τη διοργάνωση μαζί με την Οικονομική Νομισματική Επιτροπή, την κοινή αυτή συνεδρίαση. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που απεδέχθη την πρόσκλησή μας να παρίσταται. Όχι να προχωρήσει σε λεπτομέρειες όσον αφορά το επικείμενο πακέτο για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά περιμένουμε να δούμε ποιες ενδείξεις θα μας δώσει όσον αφορά το περιεχόμενο του πακέτου. Είναι σημαντικά θέματα αυτά. Και η καταχώρα εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, σημαντικότατη και άκρος ενδιαφέρουσα προβλέπεται η συζήτηση. Ευχαριστώ εκ νέου. Υιοθέτησε Οικονομική Επιτροπή και σχετική νομοθετική, νομοθετικού περιεχομένου έκθεση και περιμένουμε να λάβει πλήρως υπόψη αυτήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Αλέν ξανά έχει την Προεδρία. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε εσείς το λόγο για περίπου 15 λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαμασούρ, κύριε Γκουαλτιέρη, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Καταρχάς, θα ήθελα ως ήθιστε ειλικρινώς να σας εκφράσω τις ευχές μας. Ειλικρινείς και θερμές για τη νέα χρονιά το 2016 που μόλις ξεκίνησε και κατά τη διάρκεια του 2016 πιστεύω ότι θα συναντώμεθα τακτικά, εν πάση περιπτώσει αυτό θα επιθυμούσα. Βλέπω σαν σημάδι ότι ξεκινήσαμε στα πλαίσια της, ε, ξεκινήσαμε, τις εργασίες, ξεκινήσαμε τον προηγούμενο χώρο με την τάξη 1 και τις εργασίες τώρα με την τάξη 2 που είναι λίγο πολύ η ίδια επιτροπή από ό,τι καταλαβαίνω με την τάξη 1. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσω εκ νέου την κινητήρια δύναμη που αποτελεί αυτή η Επιτροπή στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης. Θέλουμε πιο δίκαια φορολόγηση, αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη. Τώρα περισσότερο ποτέ είναι ουσιαστικός άξονας ε, των δράσεών μας και συνεπώς και προφανώς αυτό ανήκει και στο χαρτοφυλάκιό μου. Είμαι επιφορτισμένος με τη φορολόγηση. Η παρουσία μου ενώπιον σας στις αρχές των εργασιών των εργασιών της TAX 2 και της νέας χρονιάς είναι μαρτυρία το ότι έχω αναλάβει πολιτική δέσμευση να κινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας επισημάνω ότι υπάρχει νέος γενικός διευθυντής, ο κύριος Κουέστ, ο οποίος... Πού είναι ο κύριος Κουέστ? Είναι παρόν ο κύριος Κουέστ. Ε, Ίσως είναι... Αποσύρω λοιπόν αυτό το σχόλιο, ο κ. Μοσκοβισή. Εστέ βέβαιος ότι τον είδα προηγουμένω. Και του έδωσα και κάποιες συμβουλές. Η πρώτη βασική ήταν να συνεργάζεται σε πλήρη διαφάνεια μαζί σας και να δώσει ε, τη δέουσα προσοχή στις εργασίες σας που δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε ικανοποιητικά αλλά θα πρέπει να παίξει τον πλήρη ρόλο του γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι καθήκον μου να σας διευκολύνω στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος. Χαιρετίζω την αποφασιστική συνεισφορά σας στην όλη προσπάθεια. Από την Επιτροπή την Οικονομική και την Επιτροπή Τάξη είναι δύο επιτροπές που διευθύνονται από δύο προέδρους που έχουν στην καρδιά τους την σωστή εκπροσώπηση στην ευρωπαϊκή στον τομέα. Το 2015 συνεργαστήκαμε στενά και θέλουμε να το κάνουμε και το 2016 και πεπισμένως θα το κάνουμε με την ίδια φιλοδοξία, επιμονή όπως και προηγουμένως. Υιοθέτησε ψηφίσματα το Ευρωκοινοβούλιο το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο πέρσι. Έπαιξαν κρίσιμο ρόλο. Ούτω ώστε να διατηρήσω εγώ την όλη πολιτική όθηση που απαιτείται και να καθορίσω τι λύσει που απαιτούνται για την ε, φόρο διαφυγή και την έλλειψη διαφάνεια που πρέπει να καταπολεμηθούν ω πραγματικότητα και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Όλοι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα που έχει δημιουργηθεί, την ορμή, την όθηση. δημιουργηθήκαν από τι εκθέσει αυτέ και από τι σχέσει. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε αποφασιστικά. Λοιπόν, τα μέτρα που προτείνεται καταδεικνύουν ότι το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συντονισμένα όσον αφορά την ανάγκη να θετηθούν μέτρα συγκεκριμένα για την πραγματική καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και να ενισχύσουμε τη φορολογική διαφάνεια. Όπως και εσείς, αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια διαφανής φορολόγηση, δίκαιη και σύγχρονη και να γίνει κανονική, να εφαρμόζεται τακτικά, να γίνει συνήθεια, το συνήθες πλαίσιο. Υπάρχουν προσδοκίες και των επιχειρήσεων και των πολιτών επ' αυτού. Υπάρχουν προσδοκίες σαφέστατες και αφορούν την δικαιοσύνη. Πρέπει οι επιχειρήσεις να ρυθμίζουν και να πληρώνουν το μερίδιο της φορολογίας τους εκεί που ε, δημιουργούν τα κέρδη τους. Είναι απλούστατο ως απέτηση. Όλα που ξεπερνούν αυτό το περιθώριο, αυτή την απέτηση, ε, δεν θα, ε, δεν θα, αν φύγω, ξεφύγουμε από αυτό, θα αποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Μια προσωπική ομολογία. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή με εξαγριώνουν. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία βολεύτηκαν στο παρελθόν διάφοροι ε, ενώ είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα και κοινωνική αδικία και οικονομική αναποτελεσματικότητα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε μαζί με την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και υπάρχουν και βασιλεύουν γιατί οι δημοσίε αρχέ δεν μπορούν να δράσουν. Ε, το συμπέρασμα ποιο είναι. Θα δράσουμε και πολύ αποφασιστικά πάνω στη μέθοδο. Ξέρω ότι είσαστε απόλυτα δεσμευμένοι πάνω σε αυτό το στόχο και εμείς και εγώ προσωπικά θα σας υποστηρίξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας πω ότι υποστηρίζω την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να συνεχίσει το έργο του. Δεσμεύομαι λοιπόν, όπως το είχα κάνει και στις συνομιλίες μας που ήταν δύσκολες αυτό το θέμα, να εξασφαλίσω την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο θεμητό δικαίωμα του Κοινοβουλίου να έχει πρόσβαση στα έγγραφα και το δικαίωμα των κρατών μελών ε, με σεβασμό των συμφωνιών και των συμφωνιών των θεσμικών οργάνων με τα κράτη. Μπαίνω τώρα στην ουσία. Καταρχάς, θα θέλω να κάνω μια μικρή ανατρομή στις δράσεις του 2015 για να σας δείξω ότι υπάρχει μια συνέπεια στις δράσεις μας και να σας δείξω ότι υπάρχει μια επιμονή των Κομισιών. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί επιθετική, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός. Έχουμε δύο βασικέ πρωτοβουλίε, ένα πακέτο για την φορολογική διαφάνεια το Μάρτιο και ένα σχέδιο δράση για την φορολογία των ε, επιχειρήσεων τον Ιούνιο του 2015. Είναι δύο πρωτοβουλίε με ευρύτατο πλαίσιο που θέτουν μία βάση για μία βαθιά μεταρρύθμιση τη ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορούμε και γρήγορα και καλά να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων παρά την στάση του Συμβουλίου, που υπάρχει εκεί μπλοκάρισμα. Ε, και εκεί η κοινή μας δράση είναι πολύ σημαντική για να κουνηθούν τα κράτη-μέλη. Και πιστεύω ότι οι τράσεις μας συνδέονται παρά τις διαφορετικές ευαισθησίες που έχουμε. Πρόκειται για κανόνες που αποτελούν δεσμεύσεις, ε, δεν μπορούν να αγνοηθούν, υπάρχουν τα κράτη-μέλη ε, Επίση, δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε την νομιμότητα του Συμβουλίου, αλλά δεν μπορεί να είναι δικαιολογία αυτή. Η υιοθέτηση τη οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά ε, τι φορολογικέ συμφωνίε το περασμένο κατα... καλοκαίρι είναι μια μεγάλη επιτυχία, το επαναλαμβάνω. Και φυσικά δεν, δεν πήγαμε τόσο μακριά όσο ήθελε η Κομισιόν και ούτε τόσο μακριά όσο επιθυμούσε το Κοινοβούλιο. Αλλά χάρη στην πολιτική πίεση που ασκήσατε, ε, το είπα στην Ολομέλεια και το επαναλαμβάνω, πετύχαμε ένα συμβιβασμό ικανοποιητικό ως προς την ποιότητά του και ανέλπιστο. Όχι σε σχέση με ό,τι συνέβαινε πριν, αλλά και σε σχέση με το τι μπορούσαμε να περιμένουμε αρχικά. Η δουλειά ε, προχωρεί με μεγάλα βήματα και σε πολλούς άλλους τομείς, σε ό,τι αφορά τις ε, τιμές μεταβίβασης, ε, σε ό,τι αφορά επίσης την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των ε, εταιριών, το CCTB στα αγγλικά, ή την μεταρρύθμιση των σχετικών οδηγιών. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Η ατζέντα της Κομισιόν του 2016 είναι βαριά. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όμως που επιβάλλουν κάποια όρια και δεν μπορώ να μιλήσω ε, ανοιχτά όσο θα ήθελα. Ε, σέβομαι αυτά τα όρια. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβετε υπόψη και εγώ τα λαμβάνω υπόψη, σεβόμενος την, την άποψη του συνόλου των επιτρόπων. Εμείς πάντως μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε τις προτάσεις. Στο τέλος του μήνα θα παρουσιάσουμε ένα φιλόδοξο πακέτο για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. Το Anti-Tax Avoidance Package θα είναι η πρώτη πράξη του προγράμματος του 2016 και ένα πακέτο το οποίο θα είναι ο κρογωνιαίος λήθος για τη δουλειά των επόμενων μηνών. Ξέρετε τον, την αφετηρία μας, δηλαδή ποια είναι η διάγνωση που έχουμε κάνει. Ε, η ιδιαιτερότητα της ενιαίας αγοράς ε, μας αναγκάζει να έχουμε συντονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και Μερικέ φορέ θα πάμε πιο μακριά από τις συστάσεις του ΟΣΑΣ ό,τι αφορά το πρόγραμμα BEPS το πακέτο ακριβώ αυτό το στόχο. Θα είναι επίση ένα συνολικό πακέτο. Συνολικό γιατί θα έχει πρωτοβουλίε νομοθετική φύσεω, αλλά και μη νομοθετικής φύσεως. Ε, συνολικό γιατί θα έχει και εσωτερική διάσταση και εξωτερική διάσταση. Θα υπάρχει μια εξωτερική στρατηγική απέναντι σε τρίτε χώρε ό,τι αφορά τα πλαίσια τη καλή ε, φορολογική διακυβέρνηση και συνολικό, γιατί θα δώσει συνέχεια στι συζητήσει ε, που έχουν γίνει ε, στα πλαίσια του Project BEPS σε διεθνές επίπεδο ε, με βάση τις εργασίες του ΩΣΑ και στα πλαίσια και τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια του G20. Όταν υιοθετηθεί από το Σώμα των Επιτρόπων θα επανέλθω στο Κοινοβούλιο για να σας το παρουσιάσω ε, εν πάση λεπτομερία. Είναι χρήσιμο νομίζω αυτό. Να μην σας κρύψω ότι η Κομισιόν έχει ξαναεπανεκκινήσει το project για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιριών και θέλω να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι αυτό το project δίνει επίσης μια συνολική λύση σε ό,τι αφορά την μεταφορά κερδών στο εσωτερικό της Ένωσης και επιτρέπει μια ε, δικαιότερη φορολογική μάχη ή φορολογικό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων. Έτσι θα υπάρξει μια αναζωγόνηση του CCTB. Ε, ούτω ώστε να φτάσουμε στην συντομότερη δυνατή συμφωνία. Θα ξεκινήσουμε με την κοινωνική ενωπημένη βάση και μετά θα φτάσουμε σε ένα πραγματικό CCTB. Θέλω να κρατήσουμε το CCC. Ξεκινάμε με την πρώτη φάση. Δεν θα σταματήσουμε στην πρώτη φάση. Θα υπάρξει δηλαδή μια συνολική προσέγγιση. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η Κομισιόν κρατάει το, το ρυθμό της ό,τι αφορά την, τις εκθέσεις αναχώρα. Ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να τελειώσουμε τις μελέτες αντικτύπου που είναι εξελίξη. Εν συνεχεία με, τον, με τους συναδέλφους, την κυρία Γιούροβα κτλ. Θα κάνουμε τα, τα απαραίτητα την επόμενη άνοιξη, ούτως ώστε να έχουμε τις απαραίτητες προτάσεις. Ε, ξέρετε ποια είναι η προσωπική μου θέση, σας την έχω πει. Θέλω να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Το έχω πει αυτό στους ε, νομοθέτε. Ε, το θέμα είναι αν βραχυπρόθεσμα θα το πετύχουμε. Θα πετύχουμε την απόλυτη διαφάνεια δηλαδή. Ή αν θα λάβουμε υπόψη ε, και κάποια προβλήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα και το συζητήσαμε με τον Αλάν Λαμασούχ στα πλαίσια να κλείσουμε τώρα οριστικά το θέμα. Κλείνω, κλείνω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει, ξεκίνησε το 2015 μια ευρεία προσπάθεια μεταρρύθμισης και θα συνεχίσουμε το 2016 με ταχύ Ε, στη Χάγη το, πήγα το Δεκέμβριο και την περασμένη εβδομάδα στο Άμστερνταμ και συζήτησα με τους Υπουργούς Οικονομικών της, των κάτω χωρών, που θα είναι και πρόεδρος στο Eurogroup. Καλό είναι αυτό. Ε, και με τον κύριο Βίπς, ε, που είναι επίσης υπουργός και θα παρακολουθήσει αυτές τις εργασίες. Και έχω την αίσθηση ότι η Προεδρία των κάτω χωρών ε, της τις φιλοδοξίες της Κομισιόν και έχει την πρόθεση να τα καταφέρει εξίσου καλά με τη Λουξεμβουργέζικη Προεδρία που ήταν ήδη θαυμάσια. Πιστεύω ότι το πακέτο BEPS ε, θα υιοθετηθεί μέχρι το τέλος ε, της ε, Ολλανδικής Προεδρίας. Αυτό θέλει και ο Ντάισεμπλουμ. Η Μάργκρετ Βάισταγκε επίσης έχει πολλές φιλοδοξίες για το θέμα των επιχειρήσεων. Το βελγικό καθεστώς των υπερβολικών κερδών είναι παράνομο. και θα ανακτήσουμε διάφορα χρήματα από διάφορες επιχειρήσεις. Για όλα αυτά τα μέτρα η Κομισιόν Juncker βασίζεται στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου και κυρίως των δύο επιτροπών σας. Η στενή μας συνεργασία είναι προϋπόθεση, θα πρέπει να συνεχιστεί γιατί συμμεριζόμαστε, είμαι πεπισμένος και το είδα αυτό. Έχουμε τους ίδιους στόχους. Θέλουμε διαφάνεια στις ε, πολυεθνικές γιατί ε, και δίνει, ανταμείβει αυτούς που παίζουν το παιχνίδι και τιμωρεί αυτούς που δεν το παίζουν σωστά. Και επίσης ε, βοηθάει στη σύγκληση των εθνικών μέτρων. Η μεταρρύθμιση του συστήματος ε, θα, μας, θα αλλάξει τις νοοτροπίες, θα αλλάξει τα μυαλά και έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. το είπα σε διάφορα φόρουμ ότι η επανάσταση αυτή με τη μεταρρύθμιση έχει ξεκινήσει και τίποτα δεν τη σταματάει. Όλοι όσοι αντιδρούν ε, απλώς ε, καθυστέρηση προκαλούν. Δεν πρέπει να κερδίσουν. Γιατί για να δημιουργηθεί πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα ε, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, το περιμένουν οι πολίτες μας με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, των θεσμικών οργάνων, των κρατών κτλ. Όλοι θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση και είμαι πεπισμένος ότι η Κομισιόν θα σας συνοδεύσει ούτω ώστε στο πλευρό σας να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και μαζί να υλοποιήσουμε με επιτυχία αυτή την πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση. Και πιστεύω ότι το 2006 θα είναι η χρονιά της φορολογικής διαφάνειας. Θα είναι η χρονιά των πετυχημένων φορολογικών μέτρων. Δεσμεύομαι γι' αυτό ενώπιόν σας. Ε, πολύ καλά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αναφερθήκατε στην Επιτροπή Φεστάγκερ, είμαστε σε επαφή μαζί της. Συνεφώνησε επί της αρχής να έρθει εδώ και να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις και να ενημερωθούμε για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε στα πλαίσια των ευθυνών που υπέχει. Έχουμε κατάλογο εντυπωσιακό ομιλητών. Θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο ρεταπαντήσεων της Επιτροπής Οικονομικής Δηλαδή θα διαθέτουμε λεπτά αναερώτηση ζητώντας από το μέλος που θα θέσει το ερώτημα να διαθέσει δύο λεπτά περίπου, τόσο ώστε να έχει επαρκή χρόνο ο Επίτροπος να απαντήσει. Πρώτος, Βάλτς, εν ονόματι του ισχυρού ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Καλή χρονιά και από μένα και από το ΕΛΚ. Ωραία αυτά τα οποία μας είπατε. Νομίζω πως μπορούμε να εργαστούμε με αυτά ως βάση φέτος και σωστά είπατε πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό της ε, Κομισιόν. Αυτή είναι και η δική μου άποψη. Γι' αυτό με χαροποίησαν αυτά τα οποία είπατε. Δύο πράγματα θα ήθελα να αναφέρω και να σταθώ σε αυτά. Πρώτον βεβαίως έχουμε τις εκθέσεις αν χώρα. Εσείς είστε υπέρ ενός στιβαρού τέτοιου συστήματος και η Κομισιόν είπε πως θα υποβάλει και μια αναλογική πρόταση. Βεβαίως μπορεί κανείς να πει πως η Κομισιόν ε, προχωρεί και πιέζει, κάτι το οποίο χαιρετίζω. Αλλά το θέμα είναι οι προτάσεις που θα φέρετε να συμβάζονται με αυτά τα οποία συζητούνται διεθνώς στον ΟΣΑ. Γι' αυτό θα με ενδιέφερε να μάθω πώς ε, θα αντιμετωπίσει η Κομισιόν τον πιθανό κίνδυνο ανταγωνιστικού μειονεκτήματος ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αν είναι δηλαδή να υποβληθούν σε αυτές ε, τις διατάξεις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά όχι επιχειρήσεις άλλων χωρών. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα μπορέσετε να διακρίνετε μεταξύ των μεγάλων ομίλων επιχειρήσεων και των διασυνοριακά δραστηριοποιούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί συζητάμε εδώ και χρόνια βεβαίω για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Θεωρώ πως η Κομισιόν θα πρέπει εδώ πέρα να επιμείνει παρά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη. Το ερώτημα λοιπόν είναι πως έχει εντός η, Κομισιόν αυτή τη στιγμή η συζήτηση για ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Μπάλτς. Χαίρομαι για αυτά που είπατε η ομάδα σας που είναι πάρα πολύ σημαντική στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλουμε να είναι διακομματική προσέγγιση. Υπάρχει συμφωνία από όλες τις πλευρές γι' αυτό. Όσον αφορά το country by country, τις εκθέσεις κατά χώρα. Εγώ υπερθεματίζω. Χρειάζεται διαφάνεια. Υπάρχει μια φετηρία, προφανής. Η ελάχιστη βάση είναι αυτή που καθορίζει τον ΩΣΑ. Θέλει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικήσεων και οι προτάσει που βάλουμε θα λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον αυτό. Ερώτηση. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια και να πάμε ω τη δημοσίευση των στοιχείων. Σχετικά με αυτό μπορώ να πω τι απόψει μου, τις σκέψει μου. Υπέρ είμαι προσωπικά, αλλά δεν θα πρέπει να θεσπίσουμε διάταξη που θα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα τις αποδυναμώνει εν συγκρίση με τους ξένους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να περιμένουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά των ξένων εταιριών, κυρίως των Αμερικανικών. Αυτό είναι ερώτημα που χρήζει απαντήσεως. Λοιπόν, θα πάρουμε μια απόφαση υπεύθυνη, σαν σώμα, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα αξίση το CCTB, θα κινηθούμε σε δύο στάδια. Μη λησμονούμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή σειρά. Δεν ολοκληρώσαμε ακόμα τις συζητήσεις όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο. Θέλουμε αποτελεσματική φορολόγηση, αυτή είναι η αρχή. Άρα καμία επιχείρηση δεν είναι αυτή που δεν θα καταβάλει φόρους ή θα καταβάλει λιγότερους φόρους. Τελικός σκοπός είναι να καταβάλουν το φόρο οι επιχειρήσεις εκεί που δημιουργούνται τα κέρδη τους. Ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές, ε, κυρία Ελίζα Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ μαζί μας. Ε, καλή χρονιά σας εύχομαι. Και ευχαριστώ που ξεκινάτε τη χρονιά παρουσιάζοντας σημαντικό θεματολόγιο και φιλόδοξο. Λοιπόν, η ερώτησή μου αφορά επίσης και την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε. Λοιπόν, πολύ συχνά ακούγονται επικρίσεις λογικές όσον αφορά τις τροποποίησεις που έκανε το Συμβούλιο στον αφορά τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και η ερώτησή μου σχετίζεται με αυτό. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε κάποιε θέσει και στην έκθεση τη επιτροπή ΤΑΞ με τεράστια πλειοψηφία υπέρ. Από πλευρά βουλευτών που εκπροσωπούν του πολίτε. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η όθηση που έδωσε το Κοινοβούλιο δεν θα εξαφανιστεί. Στη νέα αυτή φάση όπου εκεί θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις ληφθείς αποφάσεις. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Όσον αφορά την νομοθεσία αντιπέψ, e θέλαμε εμείς να ξεπεράσουμε τα όσα γίνονται στον όσα. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις θέσεις που έχουμε εκφράσει. Δεν θέλουμε όμως να παρεμποδίσουμε την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχει νέο νόμισμα και έχουμε μεγαλύτερε απαιτήσει. Υπάρχουν κείμενα που κυκλοφορούν. Κάποιοι προσανατολισμοί του Συμβουλίου. Και η ερώτησή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιοριστεί από αυτές τις πληροφορίες που διαφεύγουν από το Συμβούλιο και που αλλάζουν κάπως την σωστή αλληλουχία των μέτρων ή θα κινηθεί ελεύθερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υποβάλει προτάσεις, θα ζητήσει στήριξη του Κοινοβουλίου για να δημιουργηθεί θεματολόγιο φιλόδοξο και σωστό χρονοδιάγραμμα που θα θέτει υπεράνω όλων τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για το λόγο. Κυρία Φερέρα, ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ξεκίνησε στη Λισαβόνα η χρονιά, άρα είναι καλή χρονιά. Τώρα για να είμαι πιο σοβάρο και λιγότερο προσωπικά θα πω ότι δεν συμμερίζομαι την αυστηρότητά σας όσον αφορά τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία που εκφράσατε. Η ομοφωνία είναι μεγάλος περιορισμός. Επιβάλλεται σε όλου και σε εμά. Άρα δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε δεν υπάρχουν τα κάτι μέλη. Θα ήταν παράλογο. Το θέμα είναι μέχρι πού ε, θα προχωρήσουμε όσον αφορά το συμβιβασμό και η ποιότητα των συμβιβασμών που επετέφθη κυρίως όσον αφορά τις αποφάσεις ε, επί Λουξεμβριανής Προεδρίας είναι σε καλό επίπεδο. Τώρα ήθελε να προχωρήσει πιο πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πιο πέρα ακόμα. Αλλά δεν θα πρέπει όμως ε, να δυσανασχετούμε. Ε, θα έχουμε οδηγία όσον αφορά την αλλαγή πληροφοριών για τις αποφάσεις φορολογικές με ενδεχόμενη αναδρομικότητα ε, με πρωτοφανή αποδοτικότητα. Τώρα όσον αφορά ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των όσων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΩΣΑ. Εμείς θα προχωρήσουμε πιο πέρα από το BEPS. Ακόμα αν θα παραμείνει βάση μας το BEPS. Θα δείτε τα διάφορα στοιχεία που συζητούνται όσον αφορά το CCTB και την προσέγγιση για τρίτες χώρες που αφορούν όλος ιδιαίτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε ευρύτερο ε, πλαίσιο όσον αφορά τις αποφάσεις για τα φορολογικά τα rulings και θα προτείνουμε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, άρα πιο συστηματική ανταλλαγή και όχι αυθόρμητη ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Διότι έτσι εμποδίζονται κάπως οι μεταρρυθμίσεις και εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Ε, θα βασιστούμε σε αποφάσεις BEPS τις αποφάσεις του ΩΣΑ και τις αποφάσεις G20 αλλά θα ακολουθήσουμε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση που θα είναι και η δική μας. Ευχαριστώ πολύ για το ECR. Ο αντιπρόεδρος Μπέντ Λουκ έχει το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε τα οποία δεν ήταν όμως πολύ συγκεκριμένα όπως και οι απαντήσεις σας. Θα ήθελα να μας πείτε όταν λέτε πως είστε απογοητευμένοι από τον όγκο της φοροαποφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι αυτός ο όγκος. Μπορείτε να μας δώσετε έναν αριθμό. Κατ' εκτίμηση. Χοντρικά δηλαδή μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Γιατί τάξη μεγέθους μιλάμε. Ποιος είναι ο όγκος που υπολογίζει η Κομισιόν κατ' έτος ε, της ε, φοροαποφυγής και δεύτερον, τι άποψη έχετε, πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα μέτρα τα οποία προτείνεται ε, δεδομένης της φοροαποφυγής. Δώστε μας και εκεί πέρα ένα χοντρικό ποσοστό. Θα μιλάμε για την πρωτοβουλία της διαφάνειας. Ποιο ποσοστό της φοροαποφυγής μπορείτε να πιάσετε. Μιλάμε δηλαδή για 2%, 10%, 15%, πόσο. Δεν μου πείτε ακριβώς, το καταλαβαίνω, αλλά μια τάξη μεγέθους πάλι. Κάποια ιδέα πρέπει να έχετε. Το ίδιο και για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Τι άποψη έχετε πάλι. Χοντρικά ένα νούμερο. Μην πείτε ότι δεν μπορείτε να μου δώσετε ακριβές νούμερο, το ξέρω. Ποιο ποσοστό μπορείτε, θεωρείτε, να πιάσετε τη φοροαποφυγή μέσω τη κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, κύριε Σοπίτροπο. Ε, συγγνώμη, κύριε Λουκ. Δεν είμαι δημοσιογράφο. Δεν είμαι θεαματικό. Δεν μπορώ να σα δώσω νούμερο που κανένα δεν έχει. Ούτε καν ο ΣΑ δεν έχει μπορέσει να ποσοτικοποιήσει την απάτη. Δικαίω λέμε ότι είναι περίπλοκο το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσει κανεί μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για την φορολόγηση του εισοδήματο. Και έχουμε πολύ σημαντικέ διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε μια φορολόγηση που να είναι κοινή. Δεν έχουμε κοινή βάση φορολόγηση. Όταν θα αποκτήσουμε κοινή βάση, ενοποιημένη βάση, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και θα μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα τις εκτιμήσεις. Τα ποσά βέβαια είναι πολύ σημαντικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαστε νούμερα για να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα. Δεν μπορώ να σας δώσω ούτε καν τάξη μεγέθους. Μετρήσαμε το μέγεθος του φαινομένου, γνωρίζουμε τους μηχανισμούς ε, για να το καταπολεμήσουμε και τα κριτήρια θα πρέπει να είναι οι απαντήσεις που αναπτύσσουμε είναι οι κατάλληλε είναι αυτές που θα επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η πεποίθησή μου είναι ότι έχουμε μια φιλόδοξη ατζέντα, την πιο φιλόδοξη που είχαμε ποτέ και αν με ακούσατε προσεκτικά η ατζέντα αυτή ή αν κοιτάξετε την έκθεση της Κομισιόν Τάξ 1, της Επιτροπής Τάξ 1, είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα έχω την ευκαιρία όμως σε επόμενους μήνες να έρθω εδώ για να πω πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Να υπενθυμίσω ότι ο ΣΑ κάνει μια εκτίμηση. Ναι, έχω χρόνο ακόμα. Κύριε Μουσκοβιση, ε, δεν πιστεύω αυτά που ακούω. Δεν έχετε καμία ιδέα χοντρικά για το μέγεθος της φοροαποφυγής και δεν έχετε καμία ιδέα για το ποιο μέρος του προβλήματος μπορείτε να πιάσετε με τις πρωτοβουλίες σας. Ειλικρινά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχετε εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και δεν μπορείτε ούτε περίπου να μας πείτε το μέγεθος του προβλήματος και το τι θεωρείτε ότι θα κάνουν τα μέτρα σας. Ειλικρινά, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Δεν καταλαβαίνω την στάση σας. Δεν μπορώ να επινοήσω νούμερα που κανένας δεν έχει. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα των μηχανισμών που δημιουργούμε για να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που ξέρουμε ότι είναι πολύ διαδεδομένο. Υπάρχουν ε, διάφορα νούμερα που δίδονται ε, από διάφορες οργανώσεις, αλλά δεν υπάρχει κοινή βάση. Και ας, σταματήσουμε τώρα εδώ πέρα με αυτό το, αυτό το στυλ και ας προχωρήσουμε μαζί. Ο μίλησε για 100 δις με 200 δις παγκοσμίω. Θα πρόκειται σίγουρα για κάποια δεκάδες της εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη. Ο Πέτερ Γέζεκ τώρα από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ αυτή τη βδομάδα θα συζητήσει το θέμα της απάτης του ΦΠΑ. Ε, μιλάμε για νούμερα ε, της τάξης των 165 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά αυτό το είδος απάτης. Εσείς τι πιστεύετε, μπορούμε να βρούμε μια αποτελεσματική λύση για να καταπολεμήσουμε την απάτη στο ΦΠΑ. Εδώ έχουμε μια κοινή βάση για το ΦΠΑ. Έχουμε εκτιμήσεις γύρω σε αυτό το ποσό που είπατε. Εγώ δεν το ανέφερα γιατί δεν ήταν το θέμα της ε, και δεν είναι το αντικείμενο των εργασιών της ΤΑΞ, της Επιτροπής ΤΑΞ. Πάντως η Κομισιόν θα προσπαθήσει και θα είναι δύσκολο τα κράτη-μέλη να δεχτούν βέβαια για να φτάσουμε σε ένα οριστικό καθεστώς του ΦΠΑ. Θα παρουσιάσουμε ένα νέο πακέτο ΦΠΑ μέσα σε αυτό το εξάμεινο ε, που θα προσπαθήσουμε να, με αυτό να σταθούμε στο ύψος ε, των περιστάσεων γιατί και αυτό το φαινόμενο είναι πολύ σημαντικό και κινείται στα επίπεδα που είπατε για το ΦΠΑ θα έχουμε μία έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά και ο Φάμπιο Τομάζη. Ευχαριστώ κύριε Μοσκοβισή. Τρέψατε μου μια παρατήρηση για τις εκθέσεις αναχώρα. Ετίζω τις θέσεις που λαμβάνεται, Ο θείος μου είναι εκεί πέρα στην Ιταλία έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση και φτιάχνει παπούτσια και πραγματικά υποφέρει από την ε, κατάσταση αυτή της ε, φοροαποφυγής ε, και γι' αυτό απορώ με τους συναδέλφους που λένε πως θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και είδαμε γιατί τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία με τις τράπεζες που έχουν εξωφρενικά κέρδη και δεν ε, ε, πλήρωναν φόρους, κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε μόνο στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων αναχώρα. Τώρα, μια ερώτηση για αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι και για το, αυτό το οποίο έγινε παραδείγματος χάρη σήμερα στο αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο βλέπουμε πως ε, τα λεφτά αυτά τελικά επιστρέφονται είτε μιλάμε για το Βέλγιο είτε για το Λουξεμβούργο όταν μιλάμε δηλαδή για τις ε, παράνομες επιδοτήσεις. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε σε κάτι ανάλογο, δηλαδή την επιστροφή χρημάτων, όχι αχαιρεωστήτως καταβληθέντων αυτή τη φορά, αλλά χρημάτων που δεν έχουν κάνει εισπραχθεί λόγω των θύμητων φορολογικών πρακτικών. Κοιτάξτε, για να έχουμε συνοχή και να σεβαστούμε το χαρτοφυλάκιο και τον συνάδελφό μου, δεν μπορώ να απαντήσω στο δεύτερο αυτό σχέδιο που δεν βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο μου. Στο πρώτο Μπορώ να σας πω ότι μπορώ να έχω μια θέση προσωπική, είναι γνωστή και μπορώ απείρως να την επαναλαμβάνω. Πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ήπειρό μας. Δεν αμφισβητώ τη μελέτη συνεπιών και αντικτύπου. Από τη στιγμή θα ξέρουμε τα πορίσματα μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016 θα κάνουμε πρόταση που θα συνάδει με τη μελέτη αντικτύπου. Εν πάση περιπτώσει ε, θα πρέπει να βασιστούμε στο ελάχιστο, στην ελάχιστη βάση. Αυτό που συστήνει ο ΩΣΑ. Ανταλλαγή αυτόματη μεταξύ, ε, πληροφοριών μεταξύ δικήσεων. Κάτι που θα εξαλείψει τις καταστάσεις που αναφέρατε. Αυτό θέλουμε η μελέτη αντικτύπου, ένα, και η ισορροπία μεταξύ διαφάνειας και προστασίας των επενδύσεων είναι τα δύο κριτήρια για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Και να προσαρμοστούμε δεόντως. Θα το συζητήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι συνάδελφοί μου είναι πιο συνετοί, πιο προσεκτικοί από ό,τι εμένα ίσως, από ό,τι εγώ μάλλον, και σε άλλα θέματα υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση. Πρέπει να κινηθούμε όμως αντικειμενικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε, να κινηθούμε αντικειμενικά. Φάμπιο, ένα λεπτό έχετε ακόμα. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναρωτήσω πώς έχει η κατάσταση με την πρόσβαση στα έγγραφα για την τάξη. Δεν έχουμε δει κάποια έγγραφα τα οποία πρέπει να τα δούμε για να μην έχουμε και τάξε τρία τελικά. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πότε θα έχουμε τελικά πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει. Όσον αφορά αυτό, ήδη δώσαμε πολλά έγγραφα. Διαπιστώνεται ότι πολλά έγγραφα πρέπει να διατίθεται και κάπου ίσως κάποια λησμονήθηκαν από αυτά που έπρεπε να διατεθούν. Οι υπηρεσίε μου κάνουν τη σωστή την επαλήθευση. Να δούνε ποια έγγραφα λείπουν. Ούτω ώστε να διατεθούν στην Επιτροπή σας. Θα διαβιβάσω τις επόμενες μέρε τα έγγραφα και τις πληροφορίε των πρόεδρο Λαμασούρ. Αλλάζει η νοοτροπία και δημιουργείται μεγάλο φόρτο εργασίας δεν υπάρχει δισταγμός από την άποψή μας και αμφισβήτηση. Έχουμε κάθε πρόθεση να συνεργαστούμε ανοιχτά με την Επιτροπή για να γίνει η αναγκαία δουλειά. Σας ευχαριστώ. Θα ζητήσουμε από τον νέο Γενικό Διευθυντή που δεν μπόρεσε να παραστεί απόψε να έρθει να μας δει και να μας δώσει και όλα τα έγγραφα. Για τους πρασίνους. Σβέγκ Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και για την φιλοδοξία που μόλις επιδείξατε κύριε Επίτροπε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ναι. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοδοξία που επιδείξατε και συμφωνούμε πως το 2006 πρέπει να είναι το έτος της Ευρωπαϊκής Φορολογικής ε, Συνεργασίας και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε, αλλά όταν ε, μπαίνουμε στις λεπτομέρειες θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. Πρώτον, αυτό το οποίο είπε η Ελίζα Φερέρα, το Κοινοβούλιο στην έκθεση Tax 1 και στην έκθεση Dodge Niedermayer είχε κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις. Είπατε πως θέλετε να πάτε πέρα από τον BEPS και επίσης αναφέρατε και την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Δεν καταλαβαίνω το εξής. το φορολογικό αυτό πακέτο θα περιέχει τις ε, προτάσεις μας ή αλλιώς πότε θα καταθέσετε νέες προτάσεις που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις οποίες ε, ψηφίσαμε. Δεύτερον, ποια θα είναι ακριβώς η διαδικασία για να ακολουθήσετε τις προτάσεις μας ή να μας πείτε γιατί δεν συμφωνείτε. Για τις BEPS λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω για την πρόταση που θα δημοσιευτεί σε δύο εβδομάδες πού θα προχωρήσετε πέρα από το μοντέλο του ΩΣΑ, τι θα γίνει με τα panel boxes, την... το πραγματικό ύψος φορολογίας και τέλος για την κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων, τώρα μαθαίνουμε από τις εταιρείε πως ε, υπάρχει μια προσέγγιση ε, και μαθαίνουμε πως ε, θα εξασθενήσει λίγο το πακέτο. Ποια είναι τα κρατη λοιπόν τα οποία σας όθησαν σε αυτή τη στάση που δεν θέλατε κιόλας εσείς αρχικά. Ευχαριστώ κύριε Σωτήρος. και euh, euh, Το αντιμπεψ. Ποια σημεία θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να βελτιωθούν στις, ε, στην νομοθεσία των κρατών μελών. Πρέπει να αποφύγουμε κάποιες ε, μεταβιβάσεις ε, κερδών. Και επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τη διπλή φορολόγηση να αποφύγουμε την διάβρωση των ε, κερδών. Η βάση της διαφετηρία ε, μας είναι η BEPS. Θέλουμε να μεταφέρουμε το BEPS σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πηγαίνοντας και πιο μακριά από το BEPS, στα δύο σημεία που ανέφερα. Προηγουμένως έδωσε την εντύπωση ότι το μπερδεύω αυτό με την ενοποιημένη βάση των επιχειρήσεων. Όχι, είναι διαφορετικά πράγματα, άλλο το BEPS και άλλο το CCTB. Ε, γιατί έχουμε αυτή τη διπλή μεθοδολογία. Φυσικά, έχουμε κάποια στοιχεία φορολόγησης εδώ και πολλά χρόνια και διαπιστώσαμε ότι παρότι είχαμε θαυμάσιες προτάσεις, δεν πετύχαμε ομοφωνία στο Συμβούλιο για το θέμα του CDB, που είναι ζωτικό και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Το πιο βασικό θέμα είναι η ενοποίηση. Έχει γίνει μια θαυμάσια δουλειά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Μαριάν Τάισεν, πρώην συναδελφό σα, που έγινε συναδελφό μου. Ε, είχαμε την επιλογή ανάμεσα στο να παρουσιάσουμε την ίδια πρόταση με τα ίδια αποτελέσματα, χωρίς αμφιβολία, δηλαδή δεν θα είχαμε την ομοφωνία, ή να προσπαθήσουμε να βρούμε μια οδό που θα μα επέτρεπε να προχωρήσουμε. Και με βάση τα όσα γνωρίσαμε για τι συζητήσει του Συμβουλίου, δεν θέλω να σα πω ότι μπορούμε να αγνοήσουμε την ομοφωνία, είναι μια, ένας περιορισμός που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ε, πρώτη, επομένως έχουμε να κάνουμε τα εξής. Σε μια πρώτη φάση κοινή βάση και εν συνεχεία ενοποίηση. Η κοινή βάση θα πρέπει να είναι ε, ένα μέσο για να πείσουμε κάποια κράτη-μέλη που είναι απρόθυμα, δεν θέλω να τα, τα ονοματίσω εδώ, για να προχωρήσουμε ε, και είναι ο μόνος τρόπος, δυστυχώς, για να προχωρήσουμε. Πολλές προτάσεις είναι αντίστοιχες με τις ε, προτάσεις τη και τη ΕΚΟΝ. Ε, το Φεβρουάριο θα αποφανθεί και η Επιτροπή. Ε, συνεχίζουμε τα... πάνω στα σημεία τα οποία δεν υπάρχουν στο πακέτο του Ιανουαρίου και εν συνεχεία θα φτιάξουμε το πακέτο αντιμπέψ και εν συνεχεία το CCTB. μπορούμε να ονειρευόμαστε πολύ περισσότερα, αλλά εγώ θέλω να προχωρήσουμε βαθμιδών, γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε καθόλου. Η FDD, Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι εδώ για να απαντήσει τις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, για την αξιολόγηση του, των εκθέσεων αναχώρα. Θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Εσείς θέλετε δημόσια ε, δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών. Ναι ή όχι. Ε, υπάρχει κάποιος λόγος που μας εμποδίζει να μας απαντήσετε ξεκάθαρα. Οι προτάσεις που θα κάνετε θα είναι φιλόδοξες, αλλά σίγουρα ε, θα υπάρχουν κάτι μέλη τα οποία θα, είναι, θα έχουν αντιρρήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν φορολογική δικαιοσύνη. Επομένως θα πρέπει να πείσετε αυτά τα πρόθυμα κρατημέλη. Ε, επίσης, τις, ε, τις συνεδριάσεις αυτές δεν θα πρέπει να τις, να τις δημοσιοποιήσετε για να μπορέσουμε να πείσουμε αυτά τα κρατημέλη, γιατί αλλιώς θα συζητάμε ατέρμονα αυτά τα θέματα. Επίσης, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις οι Ιταλοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες δεν καταλαβαίνουν αυτούς τους κανόνες. Θα τους εξηγήσω ότι μια πολυεθνική ε, κάνει φοροδιαφυγή χάρη σε ένα ε, σύστημα ενός κράτους μέσα που τα, τη διευκολύνει. Και εν συνεχεία έρχεται η Κομισιόν και τιμωράει, αυ, τιμωρεί αυτή την α, πολυεθνική ε, και αναγκάζει το κράτος μέλος να επιστρέψει αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αυτά τα χρήματα να επιστρέφουν σε αυτά τα κράτη-μέλη, έτσι. Γιατί ε, τι νόημα έχει να εισπράττει η Κομισιόν αυτά τα, μέλη, αν, τα, τα, χρήματα, εάν δεν επιστρέφουν στους πολίτες αυτά. Λοιπόν, να απαντήσω στις δύο τελευταίες ερωτήσεις, για να είμαι συνεκτικός. Δεν θέλω να είμαι, και μη, να είμαι δημιουργικός απέναντί σας. Αυτό που σας λέω είναι ότι επεξεργαζόμαστε το θέμα. Και αυτά σας ανακοινώνω. Ίσως μπορώ να δώσω λεπτομέρειες της ε, καταχώρα εκθέσεις. Θέλω να συνεργάζομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν ε, βλέπω ότι υπάρχουν και διαφορές μεταξύ σας. Ε, τα θέματα της διαφάνειας της ανταγωνιστικότητας είναι αλληλένδετα τι θα κάνουμε. Θα λάβουμε αποφάσεις. Δεν θα λάβουν υπόψη το θέμα της δημοσιότητας. Θέλουμε να συντονιστούμε με τον ΩΣΑ. Γρήγορα θα δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα, 27 Ιανουαρίου, στο Σώμα των Επιτρόπων. Θα παρουσιάσουμε τα πρώτα μέτρα για να εφαρμοστούν τάχιστα. Για τη μελέτη αντικτύπου. Τι θα προσμετρήσει. Υπάρχουν επιλογές όσον αφορά τη διαφάνεια προς το κοινό. Ο ίδιος και οι ίδιοι κάνατε μία πρόταση που είναι μία από επιλογές. Βασικό ερώτημα. Πώς επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό πρέπει να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες. Και αυτό ζητούμε να το εντοπίσει η μελέτη αντικτύπου. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που προβάλλουν κάποιοι. Κίνδυνοι για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Διότι δεν θα είναι ισότιμη η όροι ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αλλοδαπών. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα της δημοσιοποίησης των πληροφοριών όσον αφορά λογιστικά και φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Άλλη οπτική γωνία. Ποια σχέση της πολιτικής αυτής με τη διεθνή προσέγγιση, κυρίως τα BEPS. Ε Αυτά θα εξετάσει η μελέτη αντιχτύπου με κάθε σοβαρότητα και αντικειμενικά. Και βάσει της μελέτης θα προτείνουμε συμπληρώσει των όσων θα προταθούν στις 27 Ιανουαρίου. Είμαι πλήρης και συγκεκριμένος στην απάντηση. Ναι, θα γίνει ένα πρώτο βήμα. Ο ΣΑ, προτάσεις ο ΣΑ προσαρμοσμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μπορούμε, θα προχωρήσουμε πιο πέρα. Η μελέτη αντιχπού και εσείς μέσω συζητήσεως θα μας επιτρέψετε να προχωρήσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. ENF. Gerolf Hannemans. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν έχετε λάβει υπόψη τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενους μήνες ε, που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο, δηλαδή το LuxLeaks το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να κινηθούμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, προς μια ομοσπονδιακή φορολογιακή ένωση και τελικά τα LuxLeaks ε, αποτελούν ε, απλά μια αφορμή για να προωθήσετε ε, αυτό το οποίο πιστεύετε με θρησκευτικό τρόπο ότι Δηλαδή όλα τα προβλήματα λύνονται μόνο με περισσότερη Ευρώπη. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν κάνατε ως ε, Γάλλος υπουργό ε, των ε, Οικονομικών. Ενώ μιλήσατε τότε στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση για 55 δισεκατομμύρια φοροδιαφυγής. Οπότε βλέπουμε πως υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των εθνικών συζητήσεων και της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ο Υπουργός μας, ο ε, Φανόβερφελντ, είπε σήμερα πως δεν θα είναι εύκολη η συζήτηση και ουσιαστικά παραδέχεται πως θα αναβληθεί ε, η όλη αυτή η υπόθεση και μας παραπέμπει σε νομική ασφάλεια και τα λοιπά. Βεβαίως, ε, το ερώτημά μου παραμένει το... Ζήτημα, το ερώτημά μου λοιπόν είναι απλές. Γιατί είναι το Βέλγιο η μόνη και η πρώτη και η μόνη μέχρι στιγμής χώρα η οποία καλείται να εφαρμόσει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για τις υπόλοιπες ε, χώρες ε, και θα πρέπει νομίζω η Κομισιόν επίσης να φροντίζει να μην υπάρχει και μια στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεύτερον, σκοπεύει το σύνολο και το σώμα των ε, επιτρόπων να προωθήσει περαιτέρω την ε, κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων και να οδηγηθούμε σε μια ομοσπονδιακή φορολογική ένωση. Σας ευχαριστώ. Κύριος Επίτροπος, κοιτάξτε είμαι περήφανος για αυτή την περίοδο της ζωής μου. Δεν θα αναφερθώ σε αυτήν. Θυμάμαι ότι ήμουν από τους τρεις υπουργού οικονομικών της Ενώσεως μαζί με τον κύριο Γκούρια θα το θυμάται, είχα υποστηρίξει τον ΠΕΠΣ και με τον Βόλφκαν Σόιμπλε. ήμουν από τους πρώτους που πρότεινα ενισχυμένη συνεργασία για έναν φόρο όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Το Βέλγιο ήταν στο πλαίσιο αυτό και άλλες χώρες και ένα πακέτο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Και τελικά αυτό φέλησε τη Γαλλία κυρίως. Με σκανδάλιζε αυτό το θέμα από παλιά, όχι μόνο τώρα που έγινε επίτροπος, όταν ήμουν πολιτικά υπεύθυνο και όταν ήμουν πολίτης με σκανδάλιζε. Ανεξαρτήτως δημοσίου καθήκοντος που εκτελούσα. Υπάρχει απόλυτη συνοχή στις δράσεις μου. Δεν θα σας διέφυγε. Και δεν σχολιάζω εγώ τις αποφάσεις κυρίας Βεστάγκερ. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το Βέλγιο. Είχαμε το Fiat στο, τη Fiat στο Λουξεμβούργο, το Starbucks στην Ολλανδία και άλλες έρευνες σε άλλες χώρες. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει η διάκριση την κυρία Βαστάγκερ και ούτε για ε, δειλία αν θέλετε. Προωθούνται όντως, οι έρευνες. Ίσως μετά να επιθυμήσετε περισσότερες έρευνες, μεγαλύτερη ομοσπονδοποίηση όσον αφορά την προσέγγιση. Αυτό μπορεί να συζητηθεί από πλευρά σας εδώ. Πρέπει να σεβόμαστε ένα κανόνα. Ότι αυτή η συνάδελφός μας, ο συνάδελφος, ο ή η επίτροπος που είναι υπεύθυνη για ανταγωνισμό θα πρέπει να μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα. Πρέπει να μπορεί να ασκεί ελεύθερα τις ευθύνες της, να κινείται ανεξάρτητα. Και ο καθένας γνωρίζει εδώ ότι η κυρία συνάδελφος κάνει καλά τη δουλειά της. Ευχαριστώ, όπως είπα, θα έχουμε τη δυνατότητα να τη συναντήσουμε τις επόμενες εβδομάδες στα πλαίσια της Επιτροπής ΤΑΚΣ. Για το δεύτερο, η δεύτερη ομάδα των ομιλητών θα δώσω την προεδρία στον πρόεδρο κ. Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέν Ντανούτα Χούμπνερ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, έχω δύο ερωτήσεις εγώ. Η μία αφορά την ψηφιακή οικονομία, γιατί φαντάζομαι πως η Κομισιόν θα θελήσει να κάνει και κάτι για τις ε, φορολογικές ε, προκλήσεις ε, της ψηφιακής οικονομίας, η οποία διαδίδεται βεβαίως ταχύτατα και θα θέσει διάφορα φορολογικά ζητήματα άμεσης και έμεσης φορολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν η Κομισιόν Όποιο είναι υπεύθυνο σε πάση περιπτώσει σκοπεύει να κάνει κάτι από αυτού τα επόμενα χρόνια. Μετά, για αυτό το οποίο είπε ο Μπορχαρτ Μπάλτ, για την ελάχιστη πραγματική φορολογία. Γιατί σήμερα από το Υπουργό Γκραμμένια μας είπε πως το άτυπο συμβούλιο συζήτησαν το θέμα και απέχουν πάρα πολύ από συνένεση. αλλά τόνισε την ανάγκη του να επανέλθουν σε αυτήν την συζήτηση. Οπότε η Κομισιόν κάποια ιδέα πρέπει να έχει για το πώς θα πρέπει να υπάρξει κάποια ελάχιστη πραγματική φορολογία. Μήπως εσείς μπορείτε να είστε κάπως πιο συγκεκριμένος επίσης στο θέμα αυτό θα μπορούσε το Συμβόλαιο να δεχτεί κάποια ενισχυμένη συνεργασία γιατί γνωρίζουμε πως ε, στον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ε, χρειάζονται χρόνια. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε κάποιους τομείς που θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο ενισχυμένης συνεργασίας. sur, euh, για την ψηφιακή οικονομία καταρχήν. Δεν ήταν απλή η συζήτηση στα πλαίσια του G20. Εγώ συμμετείχα ως, υπουργός, ως Γάλλος Υπουργός ε, Οικονομικών. Η απάντηση BEPS και το σχέδιο δράσης μας όμως ανταποκρίνεται στα, στις προκλήσεις της οικονομίας μας που είναι και ψηφιακή. Ε, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη φορολογική την, το φορολογικό σύστημα επιχειρήσεων που είχαν ένα φορολογικό σύστημα που αφορούσε μια άλλη εποχή, την βιομηχανική εποχή. Καταρχάς, για το καθεστώς ΦΠΑ. Εδώ δουλεύω με τους συναδέλφους μου και θα κάνουμε συζητήσει για το αν θα πρέπει να ασχοληθούμε ειδικά με το ψηφιακό θέμα ή θα πρέπει να βάλουμε το ψηφιακό, τη ψηφιακή διάσταση σε μια συνολικότερη προσέγγιση για το ΦΠΑ. Δεν, σας, δεν μπορώ να απαντήσω οριστικά σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τον ελάχιστο συντηλεστή. Θεωρούμε εδώ στην Κομισιόν ότι δεν έχουμε ανάγκη από έναν ελάχιστο συντελεστή για να φτάσουμε σε μια δίκαιη φορολόγηση. Αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε στην αρχή της πραγματικής φορολόγησης, της αποτελεσματικής φορολόγησης, ούτως ώστε να πληρώνουν οι επιχειρήσεις ε, τους φόρους τους. Εκεί όπου γεννιούνται τα κέρδη. Επιμένουμε σε αυτή την αρχή. Ξέρω ότι το θέμα της ελάχιστης φορολόγησης είναι τρομερά αμφιλεγόμενο θέμα που θα ανοίξει το κουτί της Πανθαόρας και θα προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Ε, παρότι σέβομαι διαφόρους συναδέλφους και της Κομισιόν και του Συμβουλίου, δεν νομίζω ότι αυτό θα πλουθεύσει τα πράγματα. Ε, σε ό,τι αφορά την ενισχυμένη συνεργασία, για το θέμα που αναφέρατε, η απάντησή μου είναι όχι, μάλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο Κοφίν, νομίζω, το θέμα αυτό. Κύριε Επίτροπε, ω ε, συντονιστής των ε, Σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή Τάξε, χαίρομαι που ήρθατε ξανά εδώ πέρα. Οι σημερινέ μου ερωτήσεις λοιπόν αναφέρονται και στην προηγούμενη συζήτησή μας και τον διάλογο. Τον Οκτώβριο πέρσι σας είχα ρωτήσει στην Ολομέλεια για το ότι σύμφωνα με τους ερευνητές ε, τους ε, Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ ε, κατάφεραν αυτοί να έχουν πρόσβαση στην, στον κώδικα συμπεριφοράς την οποία δεν είχαμε εμείς. Επίσης η Ελίζα Φερέρα και εγώ θέσαμε μια λεγόμενη ερώτηση κατά προτεραιότητα προ την Κομισιόν ακριβώ για αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμή δυστυχώ δεν είχαμε καμία απάντηση. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω και σήμερα τι ερωτήσει αυτές. Ισχύει το ότι το έγγραφο ερωτηματολόγιο διοικητικών πρακτικών απαντήσεις των κρατών μελών ε, στην μελέτη Σίμονς και Σίμονς δόθηκε σε εξωτερικούς και υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις όπου άνθρωποι εκτός της υπηρεσίας είχαν πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία δεν είχαν οι βουλευτές της Επιτροπής ε, Τάξε ή είχαν ε, πολύ περιορισμένοι. Τέτοια έγγραφα τα οποία μπορούσαμε να τα δούμε μόνο σε ένα αναγνωστήριο ή με κάποια σημεία τους μαυρισμένα. Και αν είχαν, ε, είχαμε τέτοια περιστατικά, τώρα Επιτέλους η Επιτροπή Τάξε θα αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας ε, με βάση σωστές ε, πληροφορίες. Ευχαριστώ. Euh, Στα πλαίσια της τάξη 1 επινοήσαμε μία μέθοδο. Είχαμε δύσκολες συζητήσεις με τον πρόεδρό σας που μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε λύσεις που δεν είναι ιδανικές, αλλά συνιστούν πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Είπα προηγουμένως ότι μπορεί να, υπα... να λείπουν κάποια έγγραφα. Τώρα, αν θέλετε να φτάσουμε, να έρθουμε εδώ πέρα στο γραφείο του Λαμασού με δεκάδες κιλά ε, βιβλίων. Οκ. Okay. Ε, πάντως, η Επιτροπή Τάξ 2, όπως και η Τάξ 1, θα έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Όλα. Και για την έκθεση Σίμων Σίμος ισχύει αυτό και για την ενδιάμεση έκθεση αυτής της, εκδοχή μάλλον αυτής της έκθεσης. Δεν υπάρχει άλλο περιστατικό τέτοια φύση από ό,τι ξέρω. Ε, Πάντω, εγώ δεσμεύομαι 100% να υπάρξει διαφάνεια και να αντιμετωπίσω την DAX 2 εξίσου καλά όπως και οποιοδήποτε άλλο φορέα που εκπροσωπεί τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο. Έχετε και άλλο χρόνο, αν θέλετε. Η δεύτερη μου ερώτηση, λοιπόν. Πότε θα έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Γιατί περιοριζόμαστε σε ένα εξάμεινο όπως ξέρετε. Και μια δεύτερη ερώτηση, σύντομη για τις εκθέσεις αναχώρα. Κάποιες πτυχές αναφέρθηκαν ήδη. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην διαφορά συστάσεων όσα και των συστάσεων σύμφωνα με την οδηγία CRD4 για τις τράπεζες που έχουν ήδη δημοσιευτεί. Δεν μας φαίνεται λογικό να απαιτούμε από τις επιχειρήσεις ε, πολλές και διάφορες αναφορές. Πώς θα αποφευθεί λοιπόν αυτή η ασυνέπεια. Στον αφορά την έκθεση κατά χώρα, να επαναλάβω τι κάνουμε. Θα κινηθούμε τάχιστα. Θα λάβουμε υπόψη τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου προφανώς θα αξιολογήσουμε τις επιλογές μας. Δεύτερον, για τα έγγραφα που λείπουν. Έκανα εκτίμηση και είπα τις επόμενες ημέρες. Θα καλυφθούν τα κενά όσον αφορά τα έγγραφα. Thank you. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο του κύριου Φερνάντε. Μιλήσω γαλλιστή λοιπόν. Μιλήσαμε για τα αγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θα πρέπει να διατηρηθεί. Ε, le Parlement et la Commission το έργο του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως. Είναι το 99% των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το συγκεκριμένο θέμα είναι και ερώτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα τις υπερασπιστεί. Δεν συμφωνώ προσωπικά με την εναρμόνιση των ποσοστών της φορολόγησης, αλλά εναρμόνιση της βάσεως και εναρμόνιση των διαδικασιών, της βάσης, φορολογικής βάσεως, ασχέτη γαλλιστή. Ποια είναι η άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, εάν θα πρέπει να επιληφθούν επιβριτέρου σχεδίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να συμπεριλάβουν τους νέους φόρους την φορολόγηση χρηματοστατικών συναλλαγών και την ανάγκη που υπάρχει για νέους ευφυείς ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχουμε και εμπειρογνώμονα. Τον πρόεδρό μας, τον Αλένα Λαμασούρ, μήπως θα έπρεπε να έχουμε και ευρύτερο σχέδιο για τους ιδίους πόρους κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο όλο σχέδιο και το θέμα των νέων ιδίων πόρων. Πρώτα απ' όλα σωστά έχετε θέσει την προτεραιότητα της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Υπάρχει σχέση μεταξύ πολυεθνικών και μικρομεσαίων. Θέλουμε να είναι ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού τους. Διαφάνεια θα επιτρέπει να αποφεύγουμε φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή από τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό δίνει καλύτερε ευκαιρίες στι μικρέ επιχειρήσει. Εναρμόνιση τώρα. Περίπλοκο να μιλήσουμε για φορολογική εναρμόνιση. Είναι και το θέμα της ομοφωνίας. Ο στόχος μας είναι εναρμόνιση διαδικασιών που επιτυγχάνεται μέσω κοινή βάσεως που εν συνεχεία θα πρέπει να καταλήξει στην γενικότερη ενοποίηση. Ίσως κάποιοι έχουν απογοητευτεί όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μια προσέγγιση σε δύο στάδια που μπορεί να ακολουθηθεί για να προχωρήσουμε. Τρίτο ερώτημα, που είναι διτό θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα έχει γενική υφή. Αναφερθήκατε στην ε, ειδικότητα που έχει ο κύριος Αλέν Λαμασούρ. Με το, στην ομάδα υψηλού επίπεδου με τον κύριο Μάριο Μόντι συνεργαζόμαστε. Και θα πρέπει εκεί να βρεθούν αξιόπιστες απαντήσεις. Προσωπικά υποστηρίζω ε, ιδίους πόρους, πραγματικούς ιδίους πόρους για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πρέπει να δημιουργηθούν και δυνατότητες και αποθέματα για την Ευρωζώνη. και ποια θα είναι η διάθεση μεταξύ ε, χρηματοπιστωτικών δυνατοτήτων της Ευρωζώνης με τον κοινοτικό προπολογισμό. Είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πριν το τέλος του 2015 καταλήξαμε σε κάποια θέση με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει πολιτική συμφωνία καταρχήν και καθορίζεται ένα χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Τον Ιούνιο θα πρέπει να υπάρχουν λεπτομέρειες για τη φορολόγηση των χρηματοσυντητικών συναλλαγών. Θα δημιουργηθεί αυτός ο φόρος. Υπάρχει, έχει ξεκινήσει η πορεία και είναι αμετάκλητη. Πολλές παράμετροι θα πρέπει εκ των υστέρων να συζητηθούν. Το ποσοστό του φόρους και πώς θα γίνει ο επιμερισμός αυτού. Μέχρι τώρα δεν αποφασίστηκε τίποτα μπορεί να θεωρηθεί ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σαν ένας υποψήφιος για τους νέους ιδίους πόρους, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με καθορισμό των διαφόρων παραμέτρων. Και αν καθοριστούν αυτές οι παράμετροι θα είναι μια τεράστια πολιτική επιτυχία ήδη. Ευχαριστώ. Επιτροπή ΕΚΟΝ και Επιτροπή Προπολογισμού θα συντάξουν μια κοινή έκθεση όσον αφορά τη δημιουργία χρηματοστικού δυναμικού για την Ευρωζώνη και τις κατάλληλες δημοσιονομικές διαδικασίες. Και ελπίζουμε ότι ε, αυτό θα συμβάλλει στην όλη συζήτηση για τους νέους ίδιους πόρους. Μανουέλ Μορέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή χρονιά στον Επίτροπο τον κύριο Λέκιος τον κύριο ε, Επίτροπο. Είπατε ότι ε, όσον αφορά τη φορολόγηση έχουμε κοινή προσέγγιση. Το βλέπουμε και στις εκθέσεις που ψηφίσαμε πέρσι και στις ε, διάφορες ομιλίες πολιτικής χρειάς που ακούσαμε από πλευράς Επιτρόπου που είναι εδώ παρόν. Αλλά για να προχωρήσουμε πιο πέρα, διότι νομίζω ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται μια σαφή υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, πρώτο σημείο θέλω να θίξω όσον αφορά. Λέτε ότι θέλετε να υπάρχει στενότατη συνεργασία όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα το κατάλαβα αυτό, αλλά συζητήσαμε στην ομάδα δεδολογικού κώδικα το θέμα αυτό και θυμάμαι ότι θέλαμε κάποιες εγγύσεις. Θα ήταν πολύ καλό κάτι τέτοιο συνεχεία. Δεύτερη ερώτηση και επανέρχομαι όσον αφορά τις εκθέσεις κατά χώρα. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει κυρίως διότι γίνεται συζήτηση στα πλαίσια τη αναθεωρή οδηγία για τους μετόχους του συναδέλφου Κομφεράτη και δεν καταλαβαίνω πώς ε, η διαφάνεια είναι αντίθετη με την ανταγωνιστικότητα. Δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα. Αντιθέτω, πιστεύω ότι η διαφάνεια μπορεί να δώσει ωφέλη στον αφορά την ανταγωνιστικότητα και είναι προ όφελο των Ευρωπαίων στο σύνολό του. Λοιπόν, θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Όσον αφορά την οδηγία αναθεώρηση του θέματο των μετόχων, θα πρέπει να έχουμε την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι σαφέ. Και τέλο, είπατε πολύ θαραλέω ότι είσαστε υπέρ τη δημοσιότητα στα πλαίσια των στοιχείων κατά χώρα. Θα πείσετε του συναδέλφου σα. Και αν ναι, μπορούμε να ελπίζουμε ότι όλα θα πεμπλακούν Τελευταίο ερώτημα, λιγότερο σαφής αλλά εξίσου σημαντική, επίτροπος για οικονομικά θέματα. Και σχετικά με αυτό θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση να αφορά ένα κρισίμου σημασία θέμα που αφορά το συντονισμό των οικονομικών. Το 2016 θα μπορούσε επιτέλους να είναι η χρονιά που θα εισαχθεί μία ε, προοπτική δημοσίων εσόδων ή φορολογικών εσόδων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γιατί πιστεύουμε ότι το εξάμεινο εδράζεται μόνο επί των δαπανών, αλλά ποτέ δεν μιλάμε για το βασικό θέμα, δηλαδή τα έσοδα καταπολέμηση απάτης, φοροαποφυγής, βελτιστοποίηση επιθετικής τη φορολόγησης. Και έτσι θα πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Τελευταίο σημείο, αν επιτρέπει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, μιλάμε πολύ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτό επιτυχάνεται και μέσω τη φορολόγηση, κατά τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας και υπάρχουν λύσει ενδεχομένω. Βέβαια δεν είναι στο δικό σα απόλυτα. Μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από αυτού περισσότερο. Αυτά λοιπόν και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μορέλ. Ευχαριστώ για τι ευχέ σα. Σε ό,τι αφορά το κώδικα δικοντολογία και τα, τον επιμερισμό των ε, εγγράφων, δεσμευόμαστε ε, στη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια απέναντι στα μέλη τη ε, Επιτροπή Τάξη. Πολλά έγγραφα βασίζονται σε πληροφορίε που προτείνονται από τις, που δίδονται από τις εθνικές αρχές. Είναι μια συνεισφορά πολύ σημαντική, αν θέλουμε να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις και θετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τα κράτη-μέλη και να έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί τους. Κάνουμε μια διαβούλευση αυτή τη στιγμή με αυτά και θα σας δώσουμε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής τις επόμενες εβδομάδες με σκοπό να προχωρήσουμε τον πιο πολύ. Να φτάσουμε στο τέλος, ούτε ώστε να πετύχουμε την απόλυτη ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, σας έχω πει ποια είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Ε, εγώ δεν πιστεύω ότι η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα είναι αντίθετα πράγματα. Ε, δεν θέλω να προσπαθήσω πίσω του συναδέλφου, δεν ξέρω ποια ιδεολογική προσέγγιση έχουν. Απλώ θα δούμε όλα τα αποτελέσματα τη μέτρηση αντιπτώσεων ε, επιπτώσεων και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα συμπεράσματά μα. Ε, μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να έχουν αντίθετε απόψει. Ε, και δεν είναι μυστικό, έτσι. Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν διαφορετικέ απόψει από τι δικέ μου. Αλλά τα αποτελέσματα τη μελέτη αντικτύπου θα μα κατευθύνουν. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, τη φορολόγηση, Φυσικά υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θέλουμε όμως ε, μέσα στο 2016 και ή δυνατόν αυτό το εξάμεινο να προχωρήσουμε πάρα πολύ και στα πλαίσια του ΩΣΑ το θέμα των ιδιών πόρων ε, και μάλιστα να προχωρήσουμε με πιο ε, φιλόδοξο τρόπο. Τώρα, για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Ε, το συζήτησαν και οι Γάλλοι Υπουργοί ε, και στο τελευταίο ΕΚΟΦΗΝ και στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ θα ξανασυζητηθεί ε, και θα το θέσει ο Γάλλος συνάδελφος και έχει δίκιο. Οι συζητήσεις ήταν πάρα πολύ θετικές ε, στο ΕΚΟΦΗΝ. Η Κομισιόν ήταν, είναι έτοιμη να απαντήσει όλα τα ερωτήματα του Συμβουλίου να, και να κάνει προτάσεις επί του θέματος. Γιατί όντως, ξεριζώνοντας και κόβοντας την, τις ρίζες της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα βοηθήσουμε στην εξάλληψη της τρομοκρατίας. Είναι βασικό στοιχείο Λέγεται ότι δεν είναι στο χαρτοφυλακείο μου και όμως είναι και μάλιστα θα ξοδέψω πολύ πολιτική ενέργεια τους επόμενους μήνες γιατί θεωρώ ότι είναι ε, εξόχου ε, σημασίας. Μπερτ Λούκα. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε μόλις πως οι εκθέσεις αναχώρα μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ, άρα, την δημοσίευση συγκεντρωτικών δεδομένων για τζίρο, απασχόληση, φόρους και κέρδη. Πώς οδηγεί αυτό σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεν ξέρω, μπορείτε να με διαφωτίσετε ίσως. Αλλά έχω και μία άλλη πτυχή που θεωρώ κάπως ε, σημαντικότερη. Η έκθεση Niedermayer Dodge ε, θέλει να εισαγάγει μια ευρωπαϊκή σφραγίδα ή σήμα για δίκαιη φορολογία. Δεν ξέρω αν έχει νόημα κάτι τέτοιο και αν θεωρείτε πως έχει νόημα ποιος θα κρίνει το εάν ένας φορολογούμενος ε, εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις τους και μήπως υπάρχει ο κίνδυνος μετά κάποιες επιχειρήσεις ε, να πείσουν για κάτι τέτοιο και έτσι να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε ανταγωνιστές οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν θα έχουν αυτή τη σφραγίδα του fair taxpayer. Αυτή ήταν η ερώτησή Euh, λοιπόν, καταρχάς να πω, όπως επαναλάβω, η άποψή μου δεν υπάρχει ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ διαφάνειας δημοσίευσης και ανταγωνιστικότητας. Ακούγεται και το το επιχείρημα. Αν επιβληθεί διαφάνεια σε επιχείρηση ευρωπαϊκή αλλά όχι σε μη ευρωπαϊκή, δεν είναι ισότιμες συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Δημιουργούνται επενδυτικές ευκαιρίες για τις μεν και όχι για τις δε. Αυτό πρέπει να προσμετρήσει η μελέτη αντιχτύπου. Αυτά λοιπόν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα από αυτού. Οι μηχανισμοί οικονομικοί είναι που πρέπει να αξιολογηθούν από τη μελέτη συνεπιών. Όσον αφορά το Fair Tax Payer Labor, label, συγγνώμη, ε, κάποιου που πληρώνει τους φόρους και είναι δίκαιος όσον αφορά τους φόρους. Η Επιτροπή Οικονομική στηρίζει την υποβολή εκθέσεων κατά χώρα και αυτό το είδος της σήμανσης. Και η μελέτη συνεπιών θα εξετάσει και αυτά. Τη δυνατότητα να υπάρχει ένα σύστημα σήμανσης. Να είναι μία επιλογή. Θα αποφασιστεί το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016 και τότε θα σας παρουσιάσω τα δύο στοιχεία που θίξατε. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στα θέματα ίσως διαφανείας σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Δεύτερον, όσον αφορά τη δημοσίευση, θα προχωρήσουμε πιο πέρα, θα υπάρξει σύστημα σήμανσης. Δεν αποκλείουμε τίποτα σε αυτή την ε, φάση και η μελέτη συνεπιών θα καθορίσει τι θα αποφασίσουμε. Νέινα Η Νίνα Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε και καλή χρονιά. Τρία πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, για τη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε τη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή μας ε, και η Κομισιόν. Και θεωρώ πως μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ε, συζήτηση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Ευρώπη. Ειδικά το ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα τα ΜΜΕ είπαν πως ε, κάποιες από τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες δεν πλήρωναν φόρο επιχειρήσεων. Πραγματικά υπάρχει οργή στους πολίτες για το θέμα αυτό. Οπότε εγώ αναμένω τις προτάσεις ε, που θα μας στείλετε αλλά να έχετε υπόψη το πώς θα ακουστούν και στους συμπατριώτες μου. Δεύτερον, η πρόσφατη απόφαση της ε, Κομισιόν ε, κατά του Λουξεμβούργου και του Βελγίου τώρα ε, θεωρώ πως είναι ορόσημα όμως πως θα φροντίσουμε να μην είναι απλά βαρχιπρόθεσμες νίκες αυτές οι αποφάσεις γιατί τι θα γίνει εάν ασκήσει έφεση η βελγική κυβέρνηση όπως αναμένω ότι θα γίνει και θα χρειαστεί λίγος χρόνος, μετά οι εταιρείε θα διαμαρτυρηθούν και θα πούν ότι δεν έχει νόημα να βγάλετε μία απόφαση μετά από 10 χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε αυτή την απόφαση είναι το ότι αποζημιώνει τα κράτη-μέλη που παραβίασαν τους κανόνες ε, για τις κρατικές ενισχύσεις. Ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος. Πώς θα μπορέσουν ε, τα κράτη-μέλη τους επόμενους μήνες να προχωρήσουν σε ζητήματα φορολογίας. Και τρίτον, σύντομα, το 2014 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο νομοθέτησαν για τον τομέα του ελέγχου όμως οι υποθέσεις δείχνουν πως οι εταιρείες και οι φορολογικοί τους σύμβουλοι κυρίως ε, αυτοί οδηγούν σε αυτά τα νομικά κατασκευάσματα. Πώς θα τροποποιήσουμε λοιπόν τη σχετική νομοθεσία. Τι προτείνεται να γίνει από εδώ και μπρος. Πρώτον, έχετε δίκιο για τον αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πάρα πολύ ενεργό όσον αφορά την διαφάνεια και τα BEPS. Σα το είχα πει ότι ήταν ένα από του πρώτου υπουργού που αντέδρασε θετικά στην πρωτοβουλία του ΟΣΑ. Ήμασταν μαζί με τον Βόφκαν Σόιμπλε και τον Τζόρτζ Όσμπορν και αναμένω και τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου που θεωρώ ότι θα υπάρξει ε, στο πακέτο που θα παρουσιάσουμε τον Ιανουάριο που είναι βεβαίως σύμφωνο και με τις δεσμεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σκάνδαλο όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά σε ολόκληρη την Ένωση και ελπίζω οι Βρετανικές αρχές ε, να παραμείνουν προσιλωμένες στο στόχο. Για τα άλλα ζητήματα, η Μαργαρέτ ε, ε, Verstagen και εγώ νομίζω πως έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα οι περιπτώσεις κρατικών ισχύσεων κρίνονται ξεχωριστά η καθεμία εγώ προσπαθώ να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως σεβόμαστε ο καθένας το χαρτοφυλάκιο του άλλου και υπάρχει νομίζω απόλυτη διαφάνεια. Κατά τα λοιπά πρέπει να σεβαστούμε την διαδικασία και το κράτος δικαίου. Και βέβαια είναι θεμητό οι χώρες να προσβάλλουν την απόφαση αν θεωρούν ότι αδικήθηκαν, αλλά εμείς θεωρούμε πως ε, η Κομισιόν ε, πραγματικά έχει δράσει σωστά για τους ελέγχους τώρα. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και τον κλάδο τον ελεγκτικό έτσι ώστε οι κανόνες που έχουμε υιοθετήσει να εφαρμοστούν πλήρως από τώρα μέχρι τον Ιούνιο του 2016 όταν ε, ε, ξέρετε ότι είναι η καταληκτική ημερομηνία. Και εργαζόμαστε, όπως είπα, εντατικά για να έχουμε πραγματική πρόοδο. Ευχαριστώ. Λούντε Κνίντερμαϊερ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θετικά αυτά τα οποία μας είπατε για κάποια ελάχιστη πραγματική φορολογία μετά θα πρέπει η Κομισιόν να πάει σε μια οδηγία anti-BEPS. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αν βλέπετε κάποιον τομέα στο οποίο θα έχουμε πρόβλημα για κα... επειδή έχετε κάποια ενότητα για αυτά τα οποία προτείνει ο ΩΣΑ και ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να ζητήσω δεν ε, αφορά μόνο το ζήτημα των εταιρικών φόρων. Θα πρέπει προφανώς να συλλέγουμε όλους τους φόρους. Το άλλο ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα είναι ο ΦΠΑ. Η Κομισιόν είπε πως προκαλεί στρεβλώσεις στην οικονομία και τον προϋπολογισμό. Επειδή μιλάμε για διάφορα μέτρα βελτίωσης της συλλογής του ΦΠΑ, να αν έχετε κάποια προτίμηση για το προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάνε οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Μιλάμε για ζητήματα διασυνοριακά, ψηφιακής οικονομίας, αντιστροφής της χρέωσης ή να συνεργαστούμε αποτελεσματικότερα μέσω του να αντιπαραβάλλουμε τιμολόγια. Δεν ξέρω λοιπόν τι μπορούμε να περιμένουμε, να περιμένουμε από την Κομισιόν και πότε. Για το θέμα του πακέτου καταπολέμησης της απάτης ε, το anti-BEPS το λεγόμενο. Ε, είναι δύσκολο βεβαίω πάντα να επιτύχουμε ομοφωνία για τα φορολογικά, αλλά για αυτό το κομμάτι των προτάσεών μας ε, έχουμε μεγάλες ελπίδες γιατί το έχουμε ήδη επεξεργαστεί στο πλαίσιο του ΟΣΑ, των G20 και στο υπουργικό επίπεδο και στο επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Θεωρώ λοιπόν πως εντάξει δεν θα είναι εύκολο αλλά θα είναι δυνατό να επιτύχουμε μια συμφωνία και ελπίζω και κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Ε, το έχω συζητήσει με τον κύριο Ντάισελμπλουμ, όπως σας είπα και πριν από λίγες ημέρες. Και πριν από τις διακοπές. Θεωρώ πως έχουμε αυτή τη φιλοδοξία που θα καρποφορήσει. Άλλες προτάσεις θα είναι πιο δύσκολες η πρόταση για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Μια πρόταση η οποία δεν έχει ομόφωνη στήριξη. Και φοβάμαι πως θα συνεχίσει να είναι δύσκολη όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Κοιτάξτε, δεν είναι στο πλαίσιο της σημερινής μας συζήτησης, αλλά όπως είπα, η δεύτερη βασική μου πρόταση με το πακέτο κατά της φοροαποφυγής θα είναι μια πρόταση για μεταρρύθμιση του ΦΠΑ που θα είναι ως το δυνατόν πιο φιλόδοξη. Εδώ πέρα λοιπόν το δουλεύουμε ακόμα το ζήτημα και σκοπεύω να το συζητήσουμε το Μάρτιο. Εάν θέλετε και εσείς βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας να έρθω να το συζητήσουμε πιο λεπτομερώς αλλά βεβαίως γνωρίζω πως θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι συνολική, παγκόσμια και φιλόδοξη. Μάικλ Τόιερ. Είναι και τα γενέθλιά σας σήμερα. Όχι σήμερα, αύριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, για τις ευχές. Καλή χρονιά στους συναδέλφους και σας ευχαριστώ κύριε Μοσκοβησί για την ευκαιρία που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είπαμε πως η πρόσβαση ε, στα έγγραφα θα πρέπει τώρα να είναι δυνατή. Ως συνεισηγητής της τάξε θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ήταν δύσκολο το ότι περιμέναμε τόσο πολύ και είχαμε τόσες σελίδες ε, τυπωμένες ε, και είχαμε την εντύπωση πως ε, πέρα από αυτά τα ζητήματα των tax rulings και της φοροαποφυγής ήταν και άλλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούσαν. Τώρα, τι μπορείτε να μας πείτε για τη λεγόμενη υβριδική χρηματοδότηση για, η οποία προβλέπει παραδείγματο χάρη ε, δάνεια στα οποία, τα οποία συμμετέχουν και στο κέρδος. Θεωρείτε πως θα πρέπει να υπάρξει η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά. Ανακοινώθηκε μια πρόταση για το τέλος του μήνα. Είναι απέτηση του Κοινοβουλίου βεβαίως και έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις για δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό. Τα παρουσιάσατε τα πράγματα κάπως θετικά, αλλά η Κομισιόν εδώ πέρα δεν έχει απαντήσει στο συγκεκριμένο μου ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτό το οποίο νομοθετήσαμε, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, θα λειτουργήσει όντως. Γιατί βλέπω εδώ πέρα πως ε, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να το εξασθενήσουν αυτό. Συμφωνώ, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά βλέπουμε πως δεν λειτουργήσε η εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών. Οπότε το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να επαναληφθεί το ίδιο στο μέλλον. Μια δεύτερη ερώτηση. Έχουμε τον πρόεδρο Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο. Ο κύριος Τίμερμανς είναι από την Ολλανδία ο αντιπρόεδρος. Χώρες οι οποίες στο παρελθόν ε, είχαν ακουστεί και συνδεθεί με κάποιες ρυθμίσεις φορολογικές και με Σήμερα ο υπουργό Γκρεμένια μας είπε πως η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου προσπάθησε να συμβάλλει σε μια λύση. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι πως εσείς αισθάνεστε ότι σας υποστηρίζει ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Κομισιόν επαρκώς γιατί οι απαντήσεις μέχρι τώρα ήταν ανεπαρκείς και βεβαίως ε, είναι σαφές ότι αν η Κομισιόν δεν ορίσει ένα άτομο ε, υπεύθυνο θα προσκρούσει στην αντίσταση των κρατών μελών. Χρόνια πολλά. Σας τα λέω εκ των προτέρων. Για το ερώτημα που ναι. σας θέτω για τα υβρίδια, ναι, σε ό,τι αφορά τα Patent Box ε, συνεχίζουμε ε, τη συζήτηση στα πλαίσια του κώδικα διοντολογίας. Και αν υπάρχουν ακόμα κράτη-μέλη, τόσο το καλύτερο. Θα έχουμε μία νομοθετική, μία μη νομοθετική προσέγγιση. Αν δεν μπορέσουμε θα περάσουμε σε νομοθετική προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, γίνεται αυτόματα. Και όλη η διαφορά είναι εκεί, στο αυτόματο. Ε, και η εγγύηση είναι εξή προσπάθησα πάρα πολύ να συμμετάσχει και η Επιτροπή σε όλα αυτά. Ε, στα πλαίσια της συζήτησης κάποια κράτη-μέλη προσπάθησαν να μας βάλουν στην πάντα. Και δεν υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ δεν είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στο να ε, ανταλλάσσουν οι εθνικέ διοικήσει μόνο τις πληροφορίε. Θέλω να είναι παρούσα και η Κομισιόν, τόσο ώστε τα κράτη-μέλη να παίζουν, να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους, να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους και επίσης να υπάρχει και συνέχεια. Ε, Έρευνε, διώξει κτλ. Ε, επίσης, νομίζω ότι έχουμε μία νομοθεσία ε, που είναι καλός συμβασμός. Ε, όπως και εσείς και εγώ ήθελα να πάμε πιο μακριά, αλλά και αυτό που έχουμε δεν είναι κακό. Σε ό,τι αφορά την τελευταία σας ερώτηση. Ε, η Προεδρία του Λουξεμβούργου καταρχάς ε, πέτυχε καλά αποτελέσματα. Ήταν πολύ φιλόδοξη και συνεργάστηκα θαυμάσια με τον Πιέρ Γκαρμενιά. Ε, και επίσης είχα τη δυνατότητα ε, να πάω στην Ολλανδία για να προετοιμάσω την Ολλανδική Προεδρία. Και είμαι πεπισμένο ότι έχουν την ίδια φιλοδοξία οι κάτω χώρες και θέλουν να έχουν ε, το ίδιο καλά αποτελέσματα με το Λουξεμβούργο. Έκανα κακό αστιακή, ζητώ συγγνώμη, σε ένα άτυπο εκοφήν, όπου είπα ότι μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι οι... αυτοί που μετάνιωσαν ε... ε στην πραγματικότητα ε... είναι πιο πεπισμένοι. Θέλουν να προσπαθήσουν τόσο ώστε να αλλάξει η εικόνα της ε, Χώρα του. Και να σα πω και κάτι έτσι εμπιστευτικό. Ε, τέσμα, το έχω πει και αλλού βέβαια. Όταν έγινε επίτροπο οικονομικών και χρηματοπιστωτικών υποθέσεων, ο Γιούγκερ με έλαβε στο γραφείο του και μου είπε θα είσαι επίτροπος για τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά. Ωραία είπα. Θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε εδώ. Ε, όταν ε, έδωσα και τη συνέντευξη τύπου έμαθα εκεί τη στιγμή ότι θα είμαι και επίτροπος για τα φορολογικά. Δεν το έκανε τυχαία ο Γιούγκερ. Ήθελε αυτά τα πράγματα να συνδεθούν. Και από την άλλη ήθελε να δείξει και την πολιτική του συμπαράσταση. Ε, έχω την ε, αμέριστη στήριξή του και την στήριξη όλων των συναδέλφων. Και ομολογώ, τελευταίο κουβέντα αυτή είναι, ότι το να έχουμε μια τόσο φιλόδοξη επιτροπή τάξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεγάλο ατού. Γιατί όταν ε, υπάρχουν προθυμίες, ε, δισταγμοί κτλ. Α, σας παραπέμπω και αναφέρω το δικό σας όνομα κύριε Λαμασούρ. Και τσακ δουλεύει. Πολύ ωραία. Έχουμε και φιλοδοξία και αισιοδοξία. Καλό είναι αυτό. Χαίρομαι που έχετε αμέριστη υποστήριξη από τους συναδέλφους σας. Ε, μπορούμε να καταλήξουμε ότι η Λουξεμβουργιασική Προεδρία τα πήγε πολύ καλά και το ίδιο περιμένουμε και από τη νέα Προεδρία. Περιμένουμε την παρουσίαση του πακέτου ATP καθώς και την ε, παρουσίαση του πακέτου ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι το Φεβρουάριο θα δώσετε απαντήσεις ενώ ενώπιον της Κομισιόν ε, για την συγκεκριμένη ε, νομοθετική πρόταση που έκανε το Κοινοβούλιο, ε, που ήταν και αντικείμενο της εκθεσής μου. πολλά θα έχουμε να κάνουμε και να πούμε το 2016. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε τις πολιτικές απόψεις και την ίδια φιλοδοξία. Και τελικά λόγια είναι ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται εκεί που παράγονται και δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομική μα διακυβέρνηση εάν δεν ε, τα καταφέρουμε καλύτερα σε ό,τι αφορά την ίσπαξη των φόρων και σε ό,τι αφορά το θέμα των ιδίων πόρων. Αλλά τελευταία σαφά λόγια και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Ε, ξεκινήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της εργασίας μας το 2016. Δύο-τρεις παρατηρήσεις. Κάτι πρώτη συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Τάξη 2 μιλήσαμε για το πρόβλημα της ε, επικοινωνίας, το πρόβλημα με τα έγγραφα και σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε στο μέλλον ε, να μάθουμε εντελώς κατά τύχη ότι υπάρχει ένα καινούργιο έγγραφο το οποίο δεν είδαμε θα ήταν ε, την πρώτη φορά ο Γενικό Διευθυντής ή την επόμενη φορά ένας εκπρόσωπος της Tax να έρθει στις συνεδριάσεις μας όταν βάλουμε δηλαδή τα έγγραφα στην ημερήσια διάταξη. Ε, γιατί θα έχετε, και πιστεύω ότι θα έχετε να μας πείτε σύντομα κάτι για αυτά τα θέματα. Είπατε στα συμπεράσματά σας και είναι ένα σημείο που τόνισε ο κ. Νίτερ Μάγερ, ότι θα πρέπει να κρατήσουμε πολιτική πίεση στις κυβερνήσεις για να φτάσουμε στο τέρμα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση των προτάσεων που υπάρχουν επιτάπητος. Και η πρόταση για την αρμόνιση της ε, φορολόγησης των κερδών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το CCTB δηλαδή, ε, συντομία, να υιοθετηθούν ε, σύντομα μαζί με το σχέδιο δράσης ε, του ΟΣΑ. Θα γίνει σε δύο φάσεις βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να γίνει. Θα επανέλθετε και θα μας πείτε ότι το χρονοδιάγραμμα για το CCTB θα εξασφαλίσει ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία του χρόνου έχετε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για το πακέτο αποφυγής της φοροδιαφυγής και για το CTB. Πολλοί συνάδελφοι, ο κ. Βάλλη, η κυρία Ζήλ, ο κ. Φερνάντες, μίλησαν για το πρόβλημα των ιδίων πόρων και για την ιδιάζουσα κατάσταση που είναι η εξή. Ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάσει ένα κράτος το οποίο έδωσε μια κρατική ενίσχυση ε, μέσω φορολογίας ε, αντίθετη στις συνθήκες. Αυτό που συμβαίνει τι είναι, ότι η επιχείρηση η οποία αποφελήθηκε από την ε, κρατική ενίσχυση θα πρέπει να πληρώσει το φόρο που οφειλόταν κανονικά και ε, ποιος υποφελείται το ένοχο κράτος. Εδώ που σκεφτόμαστε το θέμα των ιδιοπόρων που θα χρηματοδοτούν τα, τον κοινοτικό προπολογισμό, αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ίσως είναι θέμα πρωτογενούς δικαίου, ίσως είναι θέμα δύσκολων πολιτικών επιλογών, ίσως πρέπει να βρούμε την κατάλληλη νομική βάση, αλλά ένα κράτος το οποίο είναι ένοχο σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού καταδικαστεί, να μην ξαναπάρει το φορολογικό αυτό έσοδο, αλλά να μέσω ε, του κοινωνικού προϋπολογισμού αυτά τα ποσά να τα να όλοι οι υπόλοιποι. Να πάνε δηλαδή αυτά τα χρήματα στο κοινοτικό προπολογισμό. Τελευταίο σημείο. Νομίζω ότι συγκλίνουν οι απόψεις, οι απόψεις για το, τις εκθέσεις ανά χώρα. Ε, αν θα είναι περιορισμέ, ε, αν θα είναι δημόσιες. Ε, το Κοινοβούλιο μέσω της ΕΚΟΝ πρότεινε να κάνουν αυτό το tax, το taxpayer label. Ε, τελικά δεν οδηγεί στο εξή, σε αυτό που θέλουν δηλαδή. Καλ, καλώντας τις επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να λειτουργήσουν, να το κάνουν. Στην Επιτροπή Τάξ ε, ήρθαν εδώ πέρα και μίλησαν κανένα δεκαπενταριά πολυεθνικές. Οι περισσότερες μεγάλες αμερικανικές ασχολούνται με την που βρίσκονται στο ψηφιακό χώρο. Ε, και αυτό που μας εντυπωσίασε είναι ότι κάποιες επιχειρήσεις είναι έτοιμες να παίξουν το παιχνίδι. Θα μπορούσαν λοιπόν να δημιουργήσουν ένα κλαμπ φίλων αυτές οι... φίλων ας πούμε της φορολογικής διαφάνειας. Και κάποιες πολυεθνικές ανακοινώνουν ότι παρότι ε, ο η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν τις υποχρεώνει ακόμα, θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους. Αυτό θα είχε θετικές επιπτώσεις και θα προωθούσε αυτές τις επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτές που δημοσιοποιούν όλα τα αποτελέσματα και κάποιες οι οποίες με την εντύπωση ότι θέλουν κάτι να κρύψουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή ΤΑΚΣ και η... θα ξανασυνδυάσουμε την Πέμπτη στις 12 και οι συντονιστές και σε αυτή την συνεδρίαση των συντονιστών θα υιοθετηθεί και το πρόγραμμα εργασίας. Ευχαριστώ και λίγη εδώ η συνεδρίαση.